Good afternoon everybody. Uh, please find... Καλησπέρα σε όλους. Παρακαλώ καθίστε. We will start this meeting. Για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Very, very soon start speak Swedish. Και πολύ πολύ σύντομα θα αρχίσω να μιλώ Σουηδικά. Βρείτε μια άδεια θέση. Eh, λοιπόν, τώρα θα τα πω σουηδικά. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Την περασμένη εβδομάδα διοργανώσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό και χαίρομαι που σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτή τη μεικτή συνεδρίαση με την Επιτροπή Γιούρε ώστε να ασχοληθούμε με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για τις επιτροπές μας. Ε, και έχουμε την πρόταση της Επιτρόπου Ρέντινγκ που εννοεί, υπονοεί ότι ο στόχος είναι να έχουμε τουλάχιστον 40% γυναίκες στα διάφορα διοικητικά συμβούλια στην Ευρώπη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο αλλά είμαι ευτυχής ε, που μπορώ να εξασφαλίσω τη συμπροεδρία μαζί με την κυρία Ρέγνερ. Και της δίνω αμέσω το λόγο. Μάλιστα, θα είμαι και εγώ σύντομη. Εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων σας εύχομαι όχι μόνο καλό απόγευμα, αλλά και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Ε, παραδοσιακά έχουμε πολύ καλή συνεργασία, η Επιτροπή δηλαδή Νομικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Γυναικών. Και επίσης Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο πρόεδρός σας, ο κύριος Γκούσταυσον, είναι εξαιρετικά συνεργάσιμος. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ, έτσι ώστε να μπούμε στην ουσία της έκθεσης, της ισόρροπης εκπροσώπησης δηλαδή των φίλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Ο λόγος πίσω στον κύριο Γκούσταυσον. Ευχαριστώ πολύ. Οι δύο συνεισηγήτριες θα αρχίσουν, θα λάβουν το λόγο. Κυρία Κράτσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία αυτή που μπορούμε σήμερα μαζί οι δύο επιτροπές που είναι υπεύθυνε για τη σύνταξη της έκθεσης αναφορικά με την οδηγία στην οποία αναφερθήκατε να βρεθούμε σήμερα μαζί διότι πράγματι το θέμα αυτό περιλαμβάνει μια πολιτική ε, εφαρμογή των αρχών, των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης που είναι η ισότητα των δύο φύλων, η ισότητα των ευκαιριών και πρόκειται όχι για μια πολιτική παρέμβαση αλλά για μια οδηγία. Οπότε η πλευρά της, νομικής, ε, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων είναι πολύ σημαντική διότι θέλουμε να προετοιμάσουμε τη βάση μιας νομοθεσίας για πρώτη φορά στο είδος αυτό, μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία θα μπορεί απρόσκοπα να βρει εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και είμαι σίγουρη να αποτελέσει και ένα παράδειγμα για άλλες περιοχές του κόσμου που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που θέλω να πω εισαγωγικά είναι ότι η πρόταση που μας έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά ευρεία και ε, προσαρμόσιμη στην ποικιλία των νομικών και των θεσμικών συστημάτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε πράγματι λοιπόν μια νομοθεσία να έχει εφαρμογή σε 27 κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, τη δική τους παράδοση στους, στους θεσμούς της αγοράς, πέρα από, την, ε, από το πολιτικό και οικονομικό σύστημα, ε, πρέπει η οδηγία να είναι αρκετά ευρεία όπως είναι η πρόταση που ήδη έχει κάνει η κυρία Ρέντινγκ. Θέλω να τονίσω ορισμένα σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για εμένα ως εισηγήτρια και πιστεύω ότι τα συμμερίζομαι και με τα μέλη της Επιτροπής. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα αυτό, λόγω της ποικιλία των καθεστώτων που υπάρχει στα διάφορα κράτη-μέλη, ε, τις, δομές των επιχειρήσεων εννοώ, αλλά και διότι είναι για πρώτη φορά που η κοινή γνώμη έρχεται αντιμέτωπη με μια τέτοια υπόθεση και πολλές φορές υπάρχουν αντιδράσεις που έχουν να κάνουν και με έλλειψη ενημέρωσης τόσο για την πρόκληση που αποτελεί αυτή η οδηγία όσο και για το, τις μεθόδους τις οποίες εισηγείται. Πολλές φορές η κοινή γνώμη νομίζει ότι θα πάρουμε εδώ μια απόφαση και αύριο πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να έχουν στα διοικητικά του συμβούλια 40% τουλάχιστον γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αναδείξουμε τις πτυχές της οδηγίας που έχουν να κάνουν με μια διαδικασία που ξεκινάει επιτέλους, ούτως ώστε οι γυναίκες να μπορούν να είναι υποψήφιες με ίσες, με ευκαιρίες όσο και ένας άνδρας στην πλαισίωση των διοικητικών συμβουλίων. Άρα η οδηγία, όπως και η ίδια η Επίτροπος λέει, δίνει έμφαση στη διαδικασία και δευτερευόντων στον υποχρεωτικό στόχο του 40% το 2020. Για μένα είναι ένα κρίσιμο σημείο αυτό. Όχι μόνο διότι είναι η ουσία της οδηγίας, όπως επαναλαμβάνω και η ίδια η Επίτροπος λέει, αλλά διότι το κείμενο χρειάζεται να το κάνει σαφές αυτό. Διότι αν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση οφείλει το 2020 να έχει 20% γυναίκες, ε, συγγνώμη, 40% γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και αν δεν το έχει αυτό υπόκειται σε κυρώσεις είναι ένας στόχος μη ρεαλιστικός. Διότι από το 2013 μέχρι το 2020 πρέπει να γίνουν αρκετές εκλογές διοικητικών συμβουλίων για να μπορέσουν χώρες που έχουν αυτή τη στιγμή 10%, 7% συμμετοχή να φτάσουν απρόσκοπα στο 40%. Άρα είναι κεφαλαιόδες να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία ανοιχτή, αξιοκρατική, ανωδική στους στόχους που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Και εδώ όμως χρειάζεται μια διευκρίνηση για το πώς μια ε, επιχείρηση, ε, ποια είναι τα κριτήρια αυτής της υγιούς διαδικασίας που τηρεί και δεν υπόκειται σε κυρώσεις αν δεν έχει φτάσει στο 40%. Εάν υποθέσουμε ότι καθαρά θα εκφραστεί ότι ο στόχος είναι η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης της διαδικασίας, τότε δεν έχει νόημα να λέμε ότι κάποιες εταιρείες ε, που έχουν λιγότερο από 10% προσωπικό γυναίκες, δεν, σε αυτές δεν εφαρμόζεται η οδηγία αν ο κορμός και η φιλοσοφία είναι μια αξιοκρατική και αποτελεσματική διαδικασία, τότε πρέπει αυτό να ισχύει για όλες τις εταιρείες και κάποια εταιρεία που δεν θα φτάσει 40% το 2020 θα μπορεί να αποδείξει ότι εξήλυσε όλες τις μεθόδους αλλά έφτασε στο 25, στο 35 και όχι στο 40. Είναι για μένα κεφαλαιόδες αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σαφή πρόταση. Απ' την άλλη πλευρά είναι πολύ σημαντικό να δούμε πού ακριβώς αναφέρεται η οδηγία. Στις εισηγμένες εταιρείες, είναι πολύ σημαντικό αυτό διότι οι εισηγμένες εταιρείες έχουν μια ευθύνη στην κοινωνία μεγαλύτερη από τις άλλες και επίσης τις δημόσιες εταιρείες που το κράτος είναι ε, εισηγμένες αλλά το κράτος είναι ε, πλειοψηφών μέτοχος. Εκεί μάλιστα ζητάει η οδηγία το 2018 να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε εάν ε, με το να λαμβάνουμε υπόψη μόνο τις μεγάλες εταιρείες, αν σε κάποιες χώρες που δεν έχουν μεγάλες εταιρείες πολλές, θα έχει ένα αντίκρισμα η οδηγία. Μήπως πρέπει να οριστεί ένα μέγεθος που δεν είναι οπωσδήποτε οι πολύ μεγάλες εταιρείες, διότι επαναλαμβάνω υπάρχουν χώρες που δεν θα έχουν τόσο μεγάλες εταιρείες για να μπορέσει να εφαρμοστεί η οδηγία. Για μένα λοιπόν είναι τα δύο κρίσιμα σημεία τα οποία πρέπει να διευκρινίσουμε το, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και πραγματικά ποιος είναι ο στόχος ο οποίος πρέπει να πετύχουμε και η μη επίτευξη υπόκειται στις κυρώσεις. Η διαδικασία, η αποτελεσματική και διαφανής ή το υποχρεωτικό 40%. Και επίσης το άλλο σημαντικό θέμα είναι οπωσδήποτε το οποίο προέκυψε η νομική βάση. Επαναλαμβάνω ότι δεν κάνουμε μια έκθεση σαν αυτή που κάναμε το 2011 που υπερψηφίστηκε η οποία περιείχε πολλά στοιχεία τα οποία είναι μέσα στην οδηγία σήμερα. Ήταν ένα πολιτικό μήνυμα ε, προς την κοινωνία, προς τα κράτη-μέλη, προς τους εταίρους, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πετύχαμε. Άνοιξε τη διαδικασία, βοήθησε αυτή η έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει την πρότασή της. Σήμερα επεξεργαζόμαστε μια πρόταση νόμου. Οπότε τα νομικά θέματα έχουν μεγάλη σημασία και γι' αυτό είναι ευτυχής η συνεργασία μας με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σταματάω εδώ και στη συζήτηση θα μπορούμε να πούμε και για άλλες πτυχές. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κράτσα. Πρωτού δώσω το λόγο στην άλλη συνεισηγήτρια, η οποία είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γιούρι. Θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών από μια Ένωση Γυναικών Νομικών της Εσθονίας. Καλωσορίσατε, λοιπόν. Είστε ευπρόσδεκτες εδώ. Και μάλιστα μου είπαν ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το συγκεκριμένο σημείο που θα συζητήσουμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην συνσηγήτρια κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε τους αριθμούς. Γνωρίζετε πόσο χαμηλό, πόσο εξαιρετικά χαμηλό είναι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιριών. 17% σε μη εκτελεστικά συμβούλια ή σε εποπτικά συμβούλια και 13,7% σε διοικητικά όργανα μεγάλων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Αυτό μας δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει χωρίς αμφιβολία και η κυρία Κράτσα το ανέφερε. Είναι προφανές ότι χρειάζεται να αλλάξει. Δεν ξέρω εάν αυτό έχει συμβεί σκόπιμα ή όχι, όμως αυτή είναι πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της θα έλεγα πως είναι αρκετά υπομονετική, έχει αφήσει χρονικά περιθώρια. Αυτή η συζήτηση δεν έχει αρχίσει αυτό φθόρμητα, αυτή η συζήτηση διεξάγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήδη από το 1984 και το 1996 είχαμε ήδη συστάσεις του Συμβουλίου για το ποσοστό γυναικών προς τις εταιρείες αυτές για αυτορύθμιση του ποσοστού αυτού. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι αυτή η απορρίθμιση δεν έχει πετύχει. Δεν ήταν ρεαλιστική λοιπόν αυτή η πρόταση αυτές οι εταιρείε είχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τη δυνατότητα να αλλάξουν την κατάσταση στα διοικητικά του συμβούλια. Δεν έχει γίνει όμως κάτι. Φυσικά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, λαμπρές, όπως η Γαλλία, η οποία ακολούθησε το παράδειγμα της Νορβηγίας στη συμμετοχή των γυναικών. Έχει δείξει εκπληκτικά αποτελέσματα και πραγματικά αυτό μας δείχνει πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι ένα μέτρο όταν υπάρχει θέληση. Η πρόταση της Κομισιόν θα έλεγα πως είναι αρκετά επιφυλακτική όσον αφορά τις αναλογίες προς τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι, για παράδειγμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Βέβαια, ο ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν με βρίσκει απολύτω ε, σύμφωνη. Δεν είναι απαραίτητο μια εταιρεία να είναι συγμένη στο χρηματιστήριο για να είναι μεγάλη. 50 ή 100 εργαζόμενοι σε μια εταιρεία δεν την κάνουν μικρή. Και αυτές οι εταιρείες θα μπορούσαν κάλλιστα να συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο. Επίσης, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Αναφέρονται οι εταιρείε εισηγμένε στο χρηματιστήριο και ο στόχος του 40%. Το 40% στις μη διοικητικές θέσεις. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβάνει πάρα, πολλά, πάρα πολλές δυνατότητες διεξόδου ή εξαιρέσεων. Και τώρα όσον αφορά τις κυρώσεις, αυτές. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει μεγάλη επιφυλακτικότητα όσον αφορά την διαδικασία. Δεν έχει δείξει την απαραίτητη πυγμή έτσι ώστε να πει ότι εντάξει χρειαζόμαστε αυτό το 40% τώρα θα το ρυθμίσουμε έτσι και εάν αυτό δεν εφαρμοστεί θα υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις. Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, συνθήκες στα διάφορα κρατημέλη και πώς θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους αυτού το 40% αναπερίπτωση. Να σας τονίσω ότι για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας ενδιαφέρει πολύ η νομική βάση της πρότασης αυτής. Επιπλέον, όταν ενημερωθήκαμε για την εκνομοδότηση του Συμβουλίου, αντανακλαστικά σκεφτήκαμε και αντιδράσαμε ταχύτατα. χρησιμοποίησαμε το άρθρο 37 του ε, εσωτερικού κανονισμού και αναλάβαμε πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας νομική υπηρεσία και να της ε, ζητήσουμε να γνωμοδοτήσει για το θέμα. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μία εξήμνησε την ε, προσπάθεια για αύξηση του ποσοστού εκπροσώπησης, από την άλλη όμως ήταν σε πολλά σημεία σύμφωνη και με την πρόταση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Οι αντιδράσεις λοιπόν ήταν λίγο διφορούμενες. Ωστόσο να πω ότι μετά από τις αναλύσεις της δική μας νομικής υπηρεσίας καταλήξαμε στο ότι καλώς αναλάβαμε αυτήν την πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία η οποία έχει πολιτικές συνέπειες εκτός από νομικές. Τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ήδη έχουμε καταθέσει ένα πρώτο σχέδιο. Να σας υπενθυμίσω ότι μαζί με την συνεισηγήτρια κυρία Κράτσα επιθυμούμε να τηρήσουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι εμείς πρέπει να το συζητήσουμε όχι μόνο ως Ευρωβουλευτές. Πρέπει να το συζητήσουμε όμως και σε εθνικό επίπεδο, με μεγάλο ενθουσιασμό, με μεγάλη ορμή. Στις 19 λοιπόν Ιουνίου θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε το θέμα με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι παρακαλώ συζητήστε, δράστε και τηρήστε το χρονοδιάγραμμα. Εμείς θέλουμε η ψηφοφορία πραγματικά να γίνει στην Ολομέλεια αυτού του Νοεμβρίου. Έχουμε πάρα πολλές ε, προπαρασκευαστικές εργασίες να κάνουμε, γι' αυτό σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. To the rapporteurs for different kind of opinions uh, uh, well here, and uh, I will first give the floor to Mrs. Cornelison, who is the rapporteur for the opinion on employment. Please, you have the floor. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Κράτσα, Πιστεύω πως αυτό θα οδηγήσει σε δράση πριν από το τέλος της εντολής μας ε, που δεν εγκρίνεται μόνο από εμά αλλά και από το Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει να έχουμε πραγματικά αυτό σαν στόχο για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιτύχουμε. Ειλικρινά πιστεύω πως τα όσα συνέβησαν στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα είναι καλό σήμα καλό μήνυμα για την υποστήριξή τους και πραγματικά ε, ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για διάφορες ε, συμβουλές ε, από συνδικάτα, επιχειρήσεις. Κάτι που προέκυψε λοιπόν σαφώς ήταν ότι θέλουν περισσότερο να λάβουμε υπόψη τη διαφοροποίηση μέσα στις διαδικασίες επιλογής, γιατί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζεται πολύ συγκεκριμένα ποια και πώς θα πρέπει να είναι η διαδικασία και πώς θα πρέπει να προσαρμοστεί. Στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να είμαστε, εξακολουθήσουμε με να είμαστε συγκεκριμένοι για το ποιε θα είναι οι διαδικασίες επιλογής και προσλήψεων. Ε, ναι, να προσαρμοστούν στον στόχο του 40% αλλά να αφήσουμε την συγκριτική επιλογή ως ένα από τα παραδείγματα, αλλά να αφήσουμε πολύ περισσότερη ελευθερία στα κράτη-μέλη και στις επιχειρήσεις για το ποια ακριβώς θα είναι η προσαρμογή και πώς θα γίνει. Ελπίζω πως αυτό θα βοηθήσει τουλάχιστον, έτσι νομίζω, πολλές επιχειρήσεις, αλλά και τα ίδια τα κράτη-μέλη, ώστε να μην διστάζουν τόσο πολύ και να προχωρήσουν στην έγκριση της πρότασης εάν αυτή έχει περισσότερο περιθώριο ελιγμού για τους ίδιους. Να τονίσω ε, βέβαια πως δεν πρόκειται μόνο για την επιλογή. Από τη στιγμή που έχεις διάφορους υποψηφίους που θέλεις να συγκρίνεις, υπάρχει και ένα διάστημα προηγούμενο όπου οι εγκεκριμένοι όλοι αυτοί οι επιλεγμένοι πρέπει να προσληφθούν. Πώς γίνεται αυτό, πώς προχωράμε σε αυτές τις προσλήψεις και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θέλαμε επίσης να μιλήσουμε σαφέστερα για τις υποχρεώσεις αναφοράς και επεξήγησης. Η Κομισιόν έχει στόχο συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη και τις εταιρείες που δεν κάνουν κάποια προσπάθεια. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να το ενισχύσουμε αυτό περισσότερο, ώστε οι εταιρείε που τα πηγαίνουν καλά και προοδεύουν να έχουν ε, υποχρεώσεις αναφοράς πολύ light, ενώ εκείνες που δεν προσπαθούν και δεν σημειώνουν πρόοδο θα πρέπει να εξηγήσουν, να εξηγηθούν γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος ώστε ενώ πραγματικά κάνει την προσπάθεια μια εταιρεία να προσαρμόσει τις διαδικασίες και να τα, να τα κάνει όλα σωστά, να υπάρχει κάποιος λόγος όπου επελέγει κάποιος άντρας αντί για μια γυναίκα. Ενώ εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς την οδηγία. Εάν όμως δεν υπάρχει κάποια σωστή αξιολόγηση, τότε θα πρέπει να επιβάλλεται η ε, ποινή, ας πούμε κύρωση. Νομίζω πως όντως αυτό θα πρέπει να είναι ένα μοντέλο που θα βρει σύμφωνα τα κράτη-μέλη και τις ε, επιχειρήσεις. Γι' αυτό Πραγματικά θέλω να ακούσω τις αντιδράσεις ε, σε όλα αυτά. Εμείς θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων αύριο το πρωί στην Επιτροπή Επασχόλησης και προσβλέπω σε αυτήν, αλλά προσβλέπω και στην έκθεση που θα γίνει από τους την συνεισηγητρία στην αρμόδια κατουσίαν Επιτροπή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα έχει το λόγο η κυρία Παρβανόβα ε, που είναι ε, υπεύθυνη γνωμοδότησης από την ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ στην Επιτροπή Εμκο. Προχώρησαν οι εργασίες μας. Ήδη έγινε μια παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Έγινε και πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και ενίσχυσα την πρότασή μου όσον αφορά τις αρμοδιότητες Μκο. Ανέφερα το υπάρχον ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και τις τάσεις που διαπιστώθηκαν τον τελευταίο χρόνο και τονίζεται επίσης και το ποσοστό γυναικών 70% που ελέγχουν το, τις αποφάσεις αφορά τις δαπάνες των καταναλωτών στον κόσμο. Και βάσει αυτών υποθέσεων έκανα τρεις ομάδες προτάσεων. Η πρώτη ομάδα αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τονίζει την ανάγκη περισσότερες γυναίκες να είναι σε διοικητικές θέσεις διότι έτσι μπορούν να δώσουν ευρύτερε απόψει όσον αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τι επιλογέ. Και αντικατοπτρίζεται και το 70% των γυναικών που ελέγχουν την κατανάλωση στον κόσμο και τι αποφάσει για την κατανάλωση στον κόσμο. Τονίζω και τα στατιστικά στοιχεία. Φαίνεται θετική σχέση μεταξύ ποικιλομορφία φύλων σε διοικητικό συμβούλιο και οικονομικών επιδόσεων των εταιριών και κερδών και κερδοφορία των επιχειρήσεων. Θετικό αντίκτυπο λειτουργικά και οικονομικά στον τη λειτουργία των ε, εταιριών. Δεύτερη ομάδα αφορά την ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείε και την ανάγκη που υπάρχει για νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως που η νομοθεσία αυτή να δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ανταγωνιστικές για τις επιχειρήσεις με τι συνοριακές συναλλαγές συνεκτικό αξιόπιστο νομικό πλαίσιο, για να εκμεταλλευτούν την πρόσβαση στην ενιαία αγορά οι εταιρείε και να πετυχαίνουν επαρκή οικονομικά αποτελέσματα. Τρίτη ομάδα προτάσεων βασίζεται στην οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως ε, αναφέρεται στον γυράσκοντα πληθυσμό, την έλλειψη δυνατότητα χρήσεως των, του μισού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενώσης για διοικητικές θέσεις επιχειρήσεις, που μειώνει την ανάπτυξη τη της οικονομίας μας αυτό. Και η τελευταία ομάδα τροπολογιών αφορά τα κίνητρα προς τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να προτείνουν κίνητρα ούτω τόσο οι επιχειρήσεις να πετύχουν πρόοδο και να αναφέρουν πρόοδο στον αφορά το σεβασμό της αρχής της ισότητας των φίλων στα διοικητικά του συμβούλια και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε δίκτυα επιχειρήσεων και να διαμορφώνονται και οι πολιτικές περιανθρωπίνων πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζεται ε, το γυναικείο φύλλο. Αυτά λοιπόν για τη δράση των επιχειρήσεων. Πρέπει να δοθούν κίνητρα όμως από τα κάτι μελη Αυτό θεωρούμε. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα συζητηθούν οι τροπολογίες στις 29 Μαΐου, ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ στις 30 Μαΐου. Ήδη έλαβα τροπολογίες των συναδέλφων, 66 τροπολογίες μέχρι τώρα, δεν είναι και τόσο πολλές και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε συμβιβαστικές τροπολογίες και ελπίζω ότι η Επιτροπή ΙΜΚΟ θα υποστηρίξει τελικά, θα υποστηρίξει την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να ακούσουμε τις δύο συνεισηγήτριες. Αφού ακούσαν και τις εισηγήτριες για τις και τις δύο εισηγήτριες, θα ακούσουμε τους βουλευτές. Η κυρία Νευλεντάβλοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη εισηγήτριές μας, την κυρία Ρέγνερ και την κυρία Κράτσα. Χαίρομαι που το θέμα είναι στα σωστά χέρια. Ε, υποστηρίζω τη συζήτηση που διεξάγεται στην ε, Επιτροπή μας, στις Επιτροπές μας. Είναι σημαντικό που συζητείτε το θέμα. Έχω κουβεντιάσει με πολλούς νέους το θέμα και θα πιστέψετε πόσο λανθασμένες πληροφορίες κυκλοφορούν εκεί έξω. Αν μιλάμε για τα διοικητικά συμβούλια, μιλάμε για εταιρείες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια. Ε, και η κυρία Κράτσα και άλλοι συνάδελφοι το υπογράμμισαν αυτό. Πιστεύει λοιπόν ο κόσμος ότι κοιτάξτε έχω μόνο τρεις ανθρώπους ε, στις εταιρείε μου. Ε, έχω δύο άντρες και πρέπει να έχω μια γυναίκα Οπότε αισθάνομαι τις ποσοστώσεις. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες και χαίρομαι που συζητούμε το θέμα και θα το συζητήσουμε εκτενέστερα όταν επιστρέψουμε στις χώρες μας και πρέπει να σπρώξουμε τη συζήτηση σε αυτό το θέμα. Και άλλη πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα. Στη χώρα μου θα αρκούσε αν 22 εταιρείε στη Σλοβακία άλλαζαν έστω και ένα άτομο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και τότε θα πετύχει να την ποσοστώσει. Δεν είναι και τόσο τεράστιο πρόβλημα για πολλέ εταιρείε. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα ήταν καλό να προωθήσουμε αυτό το κείμενο. Γιατί υπάρχουν ποσοστώσει, Γιατί ισχύει αυτή η κατάσταση. Σαν γυναίκες, επί σειρά ετών μπορούμε να ψηφίζουμε και πολλοί άρενες συνάδελφοι ακόμα αμφισβητούν το δικαίωμά μας αυτό. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την βελτίωση των θέσεων των γυναικών μέσω ποσοστώσεων. Κατά το παρελθόν οι ποσοστώσεις είχαν πάντα θετικά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε πρόοδο. Έχουν διεξαχθεί μελέτες που δείχνουν θετικά αποτελέσματα για, με την εισαγωγή ποσοστώσεων. Στην Παγκόσμια Τράπεζα λέει ότι σε διοικητικά συμβούλια υπάρχουν περισσότερε γυναίκε στο ειδικό του συμβούλιο, τα αποτελέσματα τα οικονομικά των εταιριών αυτών είναι καλύτερα. Άντρες και γυναίκες έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, πράγματι. Και αν συνεργαστούν, τότε όλα πηγαίνουν μια χαρά. Άλλο σημαντικό θέμα είναι κάτι που συζητούσαμε. Ο, αν θα έπρεπε να έχουμε ποσοστώσεις ή να μην έχουμε ποσοστώσεις στα διοικητικά συμβούλια. Γιατί να μην μιλάμε ε, για την ύπαρξη ε, ανδρών στα διοικητικά συμβούλια. Γιατί αμφισβητείται η αξία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια χωρίς να αμφισβητείται η ικανότητα των ανδρών να είναι στα διοικητικά συμβούλια. Πρέπει να αλλάξουν την οτροπία και την προσέγγιση. Να το δούμε πάλι από την γωνία. Αν πιστεύουμε ότι οι άντρε είναι οι μόνοι που μπορούν να αποφασίζουν σωστά, τότε θα μας πούν γυναίκες ότι δεν θέλουμε εισαγωγή ποσοστώσεων γιατί είναι ασφαλμένο κλπ. Θα ακουστούν διάφορες απόψεις. Και γι' αυτό η συζήτηση που κάνουμε είναι κάτι καλό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τροφή προσκέψη. Μπορεί ο κόσμος να το σκεφτεί. Είναι θέμα, δεν είναι, πρέπει να το αντιμετωπίσει. Εγώ είμαι υπέρ των ποσοστώσεων, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση που έχουμε μπροστά μας στο Κοινοβούλιο και εύχομαι κάθε τύχη σε εσά, του συζητήτριε, για να έχουμε επιτυχή έκβαση τη προσπάθεια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βίτ. Έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως εδώ προετοιμάζουμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό νομικά. Ακούσα την ε, εισηγήτρια των φιλελεύθερων και πραγματικά άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πώς τα κράτη-μέλη προετοιμάζονται για αυτή την οδηγία. Μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση και μεγάλη άγνοια και στα μέσα ενημέρωσης. Οι γυναίκες έχουν εξαιρετικά προσόντα. Υπάρχουν γυναίκες με εξαιρετικά προσόντα, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται και σπαταλάμε δηλαδή μια τεράστια ευκαιρία που έχουμε. Συνήθως αυτές οι μεγάλες εταιρείε δεν δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα κράτο μέλο. Και εάν τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικού κανόνες όσον αφορά την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, αυτό ενδεχομένω να οδηγούσε σε περιπτώσεις όπου διαφέρουν οι αναλογίες ανά κράτος μέλος και αυτό ενδεχομένω μπορεί να προκαλέσει εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Αυτό κατακαιρματίζει το νομικό πλαίσιο και εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου διαφάνεια ως προς την διαδικασία επιλογής. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο. Ήδη ανέφερα τα αποτελέσματα στην οικονομία, τις επιπτώσεις. Το γεγονός όμως ότι δεν υπάρχει καθόλου διαφάνεια είναι κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στη σταδιοδρομία των ανθρώπων αυτών, αλλά και στην ελευθερία κίνησης. Οι επενδυτές δεν εμπιστεύονται λοιπόν μια τέτοια εταιρεία. Και αυτά είναι δύο πράγματα που ήθελα να αναφέρω σχετικά με την οδηγία. Είμαι σίγουρη πως υπάρχουν πάρα πολλά, όμως μακροπρόθεσμα μας επηρεάζει όλους και όχι θετικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ πάρα πολύ τα όσα έγιναν και θα ήθελα να συνεχίσω βασιζόμενη στην σας. Πιστεύω πως τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν αυτό το μήνυμα στα σοβαρά. Έχω την αίσθηση ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ισορροπημένη. Δεν νομίζω όμως πως είναι τόσο τέλεια ώστε δεν χρειάζεται καθόλου βελτίωση. Και είμαι σίγουρη πως αυτή εδώ η Επιτροπή θα λάβει τα πάντα υπόψη της. Θα εξετάσει προσεκτικά την πρόταση, λέξη προς λέξη. Και θα ήθελα να πω ότι εκτός από τα κράτη-μέλη. Και εμείς πρέπει να πάρουμε την πρόταση αυτή στα σοβαρά. Διότι, εάν μπούμε στον πειρασμό να ενεργήσουμε προσωπικά και να πω ότι δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι οι συγγήτριές μας θα έχουν αυτόν τον πειρασμό. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει και πραγματικά θα ήμουν εξαιρετικά δυστυχής εάν καταλήξει αυτή η πρόταση σε αδιέξοδο, εάν δηλαδή αντί να κοιτάξουμε την ουσία, να παρουσιαστούν προβλήματα από εμάς, έτσι ώστε η έκθεση να μην γίνει δεκτή. Εάν δηλαδή κάνουμε τόσες πολλές προσθήκες, κινδυνεύουμε να συμβεί αυτό. Ενδεχομένω όχι στην Ολομέλεια, στο Συμβούλιο όμω, Εκεί θα έχουμε πολλές αντιστάσεις και αντιδράσεις. Ξέρετε τι εννοώ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα σκοτώσει την πρόταση και θα την αφήσει χαμένη για δεκαετίες. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα όλους τους συναδέλφους να τους ζητήσω μάλλον να πάρουν το ζήτημα στα σοβαρά, αλλά να είναι ρεαλιστές, πραγματιστές, διότι ε, ξέρω ότι έχουμε ενθουσιασμό, ίσως περισσότερο από ότι σε άλλες εκθέσεις, σε άλλες περιπτώσεις. Παρακαλώ όμως να μην ξεχνάμε ότι εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσετε την έκθεση αυτή στη γη, είμαστε πραγματιστές, να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε και τι είναι αδύνατο να επιτύχουμε. Μπορούμε να το συζητούμε αυτό και τις λεπτομέρειες όσο θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις στην πρόταση, σίγουρα. Ας έχουμε όμως πάντοτε υπόψη το ότι η πρόταση αυτή πρέπει να παραμείνει ρεαλιστική. Έχουμε μικρά περιθώρια αποκλήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λίχτενμπεργκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω έρθει από την Επιτροπή Μεταφορών γιατί το θέμα αυτό είναι τόσο σημαντικό. Ακριβώς γι' αυτό. Και φυσικά η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εργάζεται σκληρά γι' αυτό. Οι συνάδελφοί μου ανέφεραν ήδη τους ε, πιο σημαντικούς ε, παράγοντες. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ορισμένα σημεία τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Σημαντικά έτσι ώστε εμείς να διευκολύνουμε τη δρομολόγηση της διαδικασίας εδώ στο Κοινοβούλιο, να μπορέσουμε να είμαστε πολύ ακριβείς όπως για παράδειγμα στις ε, λεπτομέρειες, στην ε, ταξινόμηση. Οι λεπτομέρειες της ταξινόμησης στο πεδίο εφαρμογής είναι κάτι που θεωρώ πάρα πολύ ε, σημαντικό. Επίσης, η ακριβής περιγραφή της διαδικασίας επιλογής. Αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά Ίσως έχετε ήδη παρακολουθήσει τις συζητήσεις που έγιναν σε εθνικά επίπεδο για την πρόταση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι εμείς εδώ μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ τη συζήτηση πάρα πολύ σημαντική. Και πιστεύω πως Η συζήτηση μέχρι τώρα μας δείχνει ότι δεν θα μείνει πάνω από τη ζώνη το επίπεδο των συζητήσεων, ενδεχομένω να έχουμε και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί, έτσι ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή και τι ενδεχόμενε εξαιρέσει, πιστεύω πω εκεί πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί, να είμαστε σαφέστατοι έτσι ώστε να προσέξουμε να μην να επικεντρωθούμε μάλλον στα σημαντικότερα και να μην αναφερθούμε σε πράγματα που ενδεχομένως δεν χρειάζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κόντεκ να λάβει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες και τους ευρωβουλευτές για τις εκφραστήσεις απόψεις να σχολιάσω κάποιες πτυχές θα ήθελα καταρχάς όσον αφορά τη φιλικότητα της πρώτης προς επιχειρήσεις ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προετοιμάζοντας την πρόταση ήταν αυτή να είναι αναλογική και φιλική προς τις επιχειρήσεις να μην επιβάλλει αυστηρές ποσοστώσεις στις εταιρείες θέτει στόχους που συνοδεύονται από υποχρεώσεις και διαδικαστικές υποχρεώσεις συνδέονται στόχοι. Φροντίσαμε επίσης να διατηρήσουμε τον ε, το χαρακτήρα που επικρατεί ο Άριστος ως στα διοικητικά συμβούλια επιλέγεται ο καλύτερος διότι ε, χρησιμοποιείται η αντίθετη περίπτωση σαν επιχείρημα κατά των ποσοστώσεων. Θέλουμε αξιοκρατική προσέγγιση λοιπόν. Προσβλέπουμε λοιπόν στην συζήτηση του πώς η πρόταση να γίνει φιλικότερη προς επιχειρήσεις και πώς το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να διευκρινίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες της πρότασης. Και ένα τελευταίο ζήτημα. Η νομική βάση, κάτι που ετέθη εδώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως επιμένει στην άποψή τη. Θεωρεί ότι η πρόταση αυτή εδράζεται επί της ορθής νομικής βάσος άρθρο 157, παράγραφος 3 που είναι η βάση για την ομοθεσία τη σχετική με την ισότητα των φύλων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το πεδίο εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν περιορίζεται στους εργαζομένους. Καλύπτει επίσης και τους αυτοαπασχολούμενους. Χρησιμοποιήθηκε για οδηγίε μέχρι τώρα που αφορούσαν τους αυτα, και κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αθετική δράση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συνήθως αυτοαπασχολούμενα άτομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο ξανά στην συνεισηγήτριες για σύντομα σχόλια πριν τελειώσει αυτή η συζήτηση. Κυρία Μπάουρ πρώτα. Θα ήθελα... Θα ήθελα να ζητήσω από τις εισηγήτριες να επανέλθουν στο θέμα της νομικής βάσης. Ποια είναι η κατάσταση τώρα και τι μπορούμε να αναμένουμε. Μα, ωραία. Πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Ρέινερ και μετά στην κυρία Κράτσα. Μάλιστα. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για όλες τις συνεισφορές σας από τους συναδέλφους. Πραγματικά τα σημείωσα όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω πως ε, έχουμε μπροστά μας μία περίοδο συνεργασίας, εξαιρετική συνεργασίας από ό,τι είδα. Τώρα όσον αφορά τη νομική βάση, να επαναλάβω αυτό που είπα νωρίτερα εμείς στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχουμε αποφασίσει σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό να χρησιμοποιήσουμε την νομική μας υπηρεσία έτσι ώστε να συνταχθεί μια έκθεση επιρρογνωμοσύνης. Η δική μας λοιπόν νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου η οποία έκθεση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την έκθεση που ήδη έχουμε της Νομικής Επιτροπής της ε, Κομισιόν, έτσι ώστε θα μπορέσουμε να αντλήσουμε λοιπόν τα συμπεράσματα όσον αφορά την πρόταση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την νομική βάση. Η έκθεση φυσικά θα έχει τις ε, κατάλληλες αναλύσεις. Θέλουμε να είμαστε προορατικοί. Και αυτό θα είμαστε. Δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε καθόλου. Πιστεύω πως σε σαφίσει όσον αφορά τη νομική βάση και συνοπτικά να σας πω ότι από εμένα τα πράγματα έχουν ως εξή. Σε αυτή την νομοθετική περίοδο θέλουμε να επιτύχουμε κάτι, θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πατήσει γκάζι, τρέχουμε, γι' αυτό βιαζόμαστε. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, τους, τις επιχειρήσεις, τους συνδέσμους επιχειρήσεων, οι οποίοι φυσικά έχουν ε, ανησυχίες, βάσιμες ανησυχίες με το, για το τι θα γίνει. Όλους λοιπόν τους ενδιαφερόμενους, όλους τους φορείς, όσους ασχολούνται με την εταιρική διακυβέρνηση να τους συμπεριλάβουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, ένα χρονοδιάγραμμα που θα μας επιτρέψει να ασχοληθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, να μιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους αλλά να φροντίσουμε σε κάθε περίπτωση να οδηγηθούμε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Κυρία Κράτσα. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Κλείνοντας τη συζήτηση αυτή ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους για το θετικό και όριμο κλίμα που αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την υπόθεση ε, είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε στα ουσιώδη, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ επιμένω ότι θέλει διευκρίνηση του σε ποια, διαδικασία υφίστανται οι επιχειρήσεις της κυρώσης. Η, όπως είπε η κυρία Ρέγνερ, όλοι μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον, όλοι πρέπει να εμπλακούν στη συζήτηση, διότι δεν είναι μόνο οι απόψεις και εμπειρίες τους πολίτη μας, είναι να τους ξεδιαλύνουμε και τους φόβους και τις απορίες και γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν επιτυχημένη και η ακρόση που ήδη τον προηγούμενο μήνα ε, ε, κάναμε και επίσης θα έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την κατεύθυνση της επικοινωνίας και της ε, ενημέρωσης η επόμενη συνάντηση με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων στις 19 Ιουνίου. Λοιπόν, πρέπει να μείνουμε στα ουσιώδη να ε, είμαστε ρεαλιστές, να έχουμε στόχο την επιτυχία και το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό. Αν είχαμε ανάγκη ένα μήνα ακόμη θα μπορούσε να τον δώσουμε αν δούμε στη διάρκεια ότι υπάρχουν προβλήματα που χρειάζονται μεγαλύτερη επικοινωνία και επεξεργασία διότι έχουμε κακές εμπειρίες από άλλες οδηγίες οι οποίες εκκρεμούν και δεν δίνουν λύσεις σε κοινωνικά θέματα είναι ώρα να φανεί ότι είμαστε έτοιμοι σαν ευρωπαϊκά όργανα να δώσουμε μια απάντηση σε ένα θέμα το οποίο άπτεται της ουσίας, της δημοκρατίας και της απόδοσης της οικονομικής. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα εργαστούμε. Ήδη ξεκίνησε μια πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών νομικών υποθέσεων και της δικής μας Επιτροπής και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουμε και θέλω να ευχαριστήσω και τις σκιώδεις εισηγήτριες αλλά και τις ε, εισηγήτριες των γνωμοδοτήσεων διότι και αυτές έχουν να δώσουν τη μάχη τους στις δικές τους επιτροπές. Μην ξεχνάμε ότι στην Ολομέλεια που θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα θα ψηφίσει όλο το Κοινοβούλιο και όχι μόνο οι δύο επιτροπές που, είναι, ε, που έχουν την ε, ευθύνη της εισήγησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thanks uh, ευχαριστώ πολύ. Ναι, μια πρία, σύντομη παρατήρηση, ανακοίνωση, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της κυρίας Ελβάνα Κοχμαρίν, που είναι η σκιώδης μας, Θέλει καταρχήν να εκφράσει την πλήρη υποστήριξη της ομάδας του Άλτε, αλλά και να καλέσει όλα τα μέλη σε μία συζήτηση κατά τη διάρκεια του πρωινού για τις προοπτικές της πολιτικής και της πρακτικής που θα γίνει αύριο το πρωί ανάμεσα στις 8.30 και τις 9.30. Όλοι είστε προσκεκλημένοι, παρακαλώ έρθετε και συνεχίσετε να πιέζετε και να βοηθάτε τις δυο υπέροχες εισηγήτριές μας. Ευχαριστώ και πριν τελειώσουμε... Θα ήθελα να ρωτήσω τη Συμπρόεδρο αν θέλει να πει κάτι ως Συμπρόεδρος τώρα. Ναι, ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ για αυτή την εξαίρετη ευκαιρία ε, συνεργασίας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλους. Ευχαριστώ τη Συμπρόεδρο για την εξαίρετη συνεργασία. Ναι, ναι, περιμένετε, δεν τέλειωσα πρέπει επίσης να σας διαβάσω μια σειρά επίσημων δηλώσεων. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συζήτηση και όσον αφορά την κοινή, το κοινό σχέδιο έκθεση στις 29 Μαΐου θα συναντήσουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια στις 19 Ιουνίου που είναι ε, στόχος για τις προ... η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 29 Ιουλίου, Ιουνίου ε, συζήτηση 9-10 Ιουλίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους.